Όχι, ε, ο κύριο ε, Κορνάρο. Ευχαριστώ πολύ που εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορώ να παρέμβω. Θα συνεχίζω στα αγγλικά και θα πω ότι είναι πολύ σκόπιμη αυτή η στιγμή πραγματικά να επανεξετάσουμε και να καταλήξουμε σε πολιτική αξιολόγηση και κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την οικονομική υποστήριξη, σύνδρομη προς την Αίγυπτο. Είναι και ε, καλή η θετική στιγμή διότι έχει μια έκθεση που ενέκρινε και κατέθεσε το ελεγκτικό συνέδριο όσον αφορά τις δράσεις μας υπό αυτά τα προγράμματα εν προσέγγιση όσον αφορά αυτή την έκθεση βλέπουμε πραγματικά να ενδυναμώνονται, να υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία στις προσπάθειες που καταβάλουμε και στον τρόπο με το οποίο πρέπει να διαχειριζόμαστε τέτοια σχέδια και ε, με αυτές τις συστάσεις ε, που μπορούμε να δώσουμε συνέχεια σε αυτές ένα ή άλλο σημείο στο κείμενο τα ε, προγράμματα, για τα προγράμματα αυτά υπάρχουν θέματα που πρέπει να τύχουν συνέχεια και δεν είναι ο τελευταίος λόγος αυτός που εκφέρεται. Για μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς βλέπουμε ως λιδία λίθο την Αίγυπτο για τα όσα θα επακολουθήσουν και αυτά τα οποία πρέπει να ε, γίνουν και αυτά τα οποία έγιναν από την ύπατη εκπρόσωπο κυρία Άστον με μεγάλη υποστήριξη και από το δικό σας σώμα από το Ευρωκοινοβούλιο μια νέα πολιτική που θα πρέπει να διασφαλιστεί ώστε να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα σε μια ολοκληρωμένη πολιτική οικονομικής και πολιτικής ανάπτυξης καταβάλλοντας μεγαλύτερες προσπάθειες να υπάρξει μια εμβάθυνση και επέκταση της δημοκρατίας ε, εκεί. Και όλα αυτά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, σε μια προσέγγιση που λέει ότι πρέπει να υλοποιούνται τα προγράμματά μας ε, με ε, συγκεκριμένη στοχοθέτηση και επικέντρωση και ανταπόκριση στην υλοποίηση των στόχων με more for more εφαρμογή. Δηλαδή να γίνονται περισσότερα και να αποκομίζονται και περισσότερα ωφέλη ε, για όλους. Εκεί όπου βρίσκεται η Αίγυπτος σήμερα στο σταυροδρόμι το ιστορικό θα λειτουργήσει ίσως λιδία λίθος για αυτή την πολιτική. Θέλω να διασφαλίσω στα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου θα εμείνουμε και θα παραμείνουμε πιστοί σε αυτές τις αρχές και αξίες. Ε, οτιδήποτε και αν συμβεί θα συνεχίσουμε να πράττουμε στο μέτρο του εφικτού α, αυτό το οποίο πρέπει να γίνεται στην Αίγυπτο. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε μια σφαιρική ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγιση όσον αφορά τα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά θέματα, ιδιαίτερα για τους πιο ευάλωτους προγράμματα και σχέδια που θα βοηθήσουν την κοινωνία των πολιτών ώστε να μπορέσει η ε, Αίγυπτος ε, σε ένα πλαίσιο δημοκρατικό και λογοδοσίας ε, και υπευθυνότητας να μπορέσει να προχωρήσει και να μπορέσει να ενδυναμωθεί και να τονωθεί και η δημοκρατική διαδικασία, ο δημοκρατισμός αλλά και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Δραστήρια λοιπόν μπορούμε να συνδράμουμε έτσι την Αίγυπτο και βρίσκονται όλα αυτά υπό επανεξέταση και υπό εξέλιξη, εμβρευστό. Και όταν θα έχουν καθοριστεί οι επιμέρους παράμετροι θα θέλαμε φυσικά να γνωρίζουμε ποιε είναι οι κατευθυντήριε γραμμές πολιτικά και από το Ευρωκοινοβούλιο και προσβλέποντας και μελλοντικά στο ε, Συμβούλιο Υπουργών ε, Εξωτερικών Υποθέσεων ε, να δούμε τι μπορεί να γίνει σε σχέση και με την επιλογή μιας αποτελεσματικής προσέγγισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης προσβλέπω στα περαιτέρω σχόλια και ερωτήσεις από πλευρά σας. Επαρκούμε σε αυτά τα σχόλια από πλευρά μου. Ευχαριστώ. Um, ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Καρν Πίξτεν, μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να παρουσιάσουμε την ειδική μας έκθεση για την Αίγυπτο σε αυτήν εδώ την Επιτροπή. Κύριος ε, στόχος του ελεγκτικού συνεδρίου είναι να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για πολιτική συζήτηση. Αυτό το επιτυγχάνουμε, σας το υπενθυμίζω, βάσει μια πολύ αυστηρής μεθοδολογίας. Όταν ξεκινάμε λοιπόν έναν έλεγχο επιδόσεων που αφορά την αποδοτικότητα την οικονομική αποδοτικότητα και σε αυτή την περίπτωση και την αποτελεσματικότητα, ξεκινάμε πάντα σε αυτό που ονομάζουμε ένα κύριο ερώτημα για τον έλεγχο. Αυτή είναι η αφετηρία και για αυτό τον έλεγχο η συνολική, η γενική ερώτηση ήταν κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά την ενίσχυση, την ευρωπαϊκή ενίσχυση για να ε, τον έλεγχο της διακυβέρνησης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ξεκίνησε ο έλεγχος το 2007, όπως γνωρίζετε όλοι, στην αρχή του ENPI και καλύπτει ουσιαστικά δύο περιόδους. Μία υπό τον πρόεδρο Μουμπάρακ και άλλη μία υπό τον πρόεδρο Μόση. Ο έλεγχος ε, βασίστηκε στα θέματα διακυβέρνησης σε αυτό το κύριο ερώτημα. Και ουσιαστικά δύο κύριου τομεί διακυβέρνηση. Πρώτον, δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα. Δεύτερον, διαχείριση των οικονομικών και η καταπολέμηση της διαφθορά. Αυτά τα θέματα αφορούσε η περίοδος από το 2007 μέχρι το Σεπτέμβριο πέρυσι. Αυτά εξετάσαμε λοιπόν και ελπίζω ότι όλα τα μέλη αυτής εδώ της διακεκριμένης επιτροπής να πρόλαβαν να κοιτάξουν το έγγραφο και σε καθένα από τα ελεγκτικά μας έγγραφα βρίσκεται το ερώτημα του ελέγχου και μετά μια σειρά παρατηρήσεων γεγονότων, ε, δεδομένων στοιχείων που βοηθούν να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις και μετά ακολουθούν τα συμπεράσματα και οι συστάσεις. Τι διαπιστώσαμε λοιπόν συμπεράναμε ότι στο συνολικά η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση δεν κατάφεραν να διαχειριστούν την ευρωπαϊκή ενίσχυση για τη βελτίωση τη διακυβέρνηση στην Αίγυπτο αποτελεσματικά. Το ερώτημα λοιπόν είναι, ή μάλλον συγγνώμη, η απάντηση είναι ότι δεν διαχειριστήκαμε σωστά τα κονδύλια που αφιερώθηκαν στην διαχείριση της διακυβέρνησης. Οι λόγοι είναι οι πολύ δύσκολες συνθήκες στην Αίγυπτο, καθώς και η απροθυμία του Πρόεδρου Μουμπάρα και του νέου ε, Πρόεδρου Μόρσε Η απροθυμία λοιπόν της Αιγυπτιακής πλευράς. Η δεύτερη αιτία είναι οι ελλείψεις ε, στον τρόπο διαχείρισης εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Μέχρι τα Αυτά είναι τα συμπεράσματα. Θα καλούσα τα μελή της παρουσίας επιτροπής να προσέξουν κάποιες συγκεκριμένες παραγράφους. Για παράδειγμα υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα παράγραφο σε σχέση με τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, η παράγραφος 47. ...60% χονδρικά της ενίσχυσης δοθήκε σε αυτό που ονομάζουν ε, ενίσχυση του προϋπολογισμού δηλαδή να βοηθηθεί η υποστήριξη ενός αποτελεσματικού ε, συστήματος διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών. Ακόμα και σήμερα όμως στην Αίγυπτο δεν υπάρχει ανεξάρτητο γραφείο εξωτερικού ελέγχου, ούτε σχετικός οργανισμός. Δεν είναι καθόλου σαφείς οι δαπάνες του στρατού, που αντιστοιχεί σε μεγάλο κομμάτι του προπολογισμού. Δεν υπάρχει καμία καθαρότητα όσον αφορά τις δαπάνες της Προεδρίας. Υπάρχουν προβλήματα με αυτά που ονομάζονται ειδικά ταμεία ύψου σχεδόν 4 δισεκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία χρόνια. Παραμένουν λοιπόν πολλά προβλήματα όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά και τη διαχείρισή τους. Αυτά τα προβλήματα κατά την απόψή μας πρέπει να αντιμετωπιστούν. Θα είμαι πολύ σύντομος τώρα για το δεύτερο σημείο που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Καθιστάτε σαφές ότι στη συνθήκη της Λισαβόνα το άρθρο 21, παραγραφός 1, καθιστάται απόλυτα καθαρό το θέμα της στήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Και στο άρθρο 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης καθιστάται επίσης σαφές ε, το ENPI και στο ENPI νομίζω στο άρθρο 28 αναφέρονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία. Εμείς τώρα κοιτώντας τα γεγονό, κοιτάμε τα γεγονότα, τα χρήματα που έχουν δοθεί και την αιρεσιμότητα. Αυτά είχα να πω για το έγγραφο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ, ευχαριστούμε κύριε Πίνξτεν. Έχω 14 εγγεγραμμένους ομιλητές στη λίστα μου. Ο καθένας τους έχει ένα μισή λεπτό. Παρακαλώ τηρήστε το χρόνο ο κύριο Αλαφράγκα πρώτο, παρακαλώ. Κύριο Αλαφράγκα, ευχαριστώ πρόεδρε. Η κατάσταση στην Αίγυπτο είναι γνωστή πιστεύω. Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την προηγούμενη Πέμπτη μια σαφή πρόταση ψηφίσματο εκφράζοντα τη θέση του και αλλάζοντα την τελευταία στιγμή την προηγούμενη πρόταση ψηφίσματο που είχαμε διαπραγματευτεί ώστε να τηρηθούμε στι νέε εξελίξει με το στατικό πραξικόπημα. Είναι σαφέ ότι το αποτέλεσμα είναι η πόλωση και η σύγκρουση Απόλυα περαιτέρω ανθρώπινων ζώων και επιταγή τώρα που είναι να αποφύγουμε, πολιτική επιταγή, επιταγή να έχουμε ακόμα μια πιο αιματηρή πολιτική σύγκρουση που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες απώλειες και μεγαλύτερη σύγχυση. Διάβασα την έκθεση και τα συμπεράσματα του μέλους του ελεγκτικού συνεδρίου για τη χώρα για το ότι η βοήθεια αυτή δεν χρησιμοποιήθηκε αποτελεσματικά. Η ερώτηση που πρέπει να διατυπωθεί εδώ είναι αν ήταν ή δεν ήταν ε, αποτελεσματική και θα θέλαμε να ήταν ε, αποτελεσματική θα μπορούσαμε ίσως να είχαμε αποφύγει μια τέτοια κατάσταση. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει μια τέτοια κατάσταση διότι δίνουμε δισεκατομμύρια στο στράτευμα, στο στρατό της Αιγύπτου και δεν καταφέραμε να αποφύγουμε αυτή, αυτό το πραξικό με αυτή την εξέλιξη. Τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με τη Task Force. Θα είμαστε σε θέση να πείσουμε τους ε, μουσουλμάνους αδερφούς να συμμετάσχουν σε μια εκλογική διαδικασία που πιθανότατα θα χάσουν την εκλογική αυτή αντιπαράθεση. Διότι βλέποντας ότι ένα τμήμα των Ισλαμιστών υποστήριξαν τη στατιωτική παρέμβαση και νομίζω ότι εδώ είναι σημαντικό αυτό το οποίο συνέβη στους δρόμους στην Αίγυπτο με τις διαδηλώσεις θα χάσουν αυτή την αντιπαράθεση. Ολοκληρώνω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρακολουθήσει αυτή την εκλογική αντιπαράθεση. Υπό οποιουσδήποτε όρου, υπό οποιασδήποτε προποθέσει, ή θα υποστηρίξουμε αυτή την εκλογική αντι... ε, διαδικασία, αν θα είναι μια δίκαια και ολοκληρωμένη εκλογική διαδικασία. Το πιο σημαντικό είναι να ασκήσει όλε τι επιρροέ και να κάνει ό,τι περνά από το χέρι τη η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποφύγουμε μια τέτοια αιματηρή σύγκρουση όπω βλέπουμε να συμβαίνει σε άλλε χώρε. Ευχαριστούμε η κυρία Γκόμες βλέπουμε ότι η δημοκρατία δεν είναι απλώς και μόνο εκλογές. Δείτε την κατάσταση στην Τουρκία. Βέβαια, οι εκλογές είναι ένα βασικό συστατικό της δημοκρατίας. Προερχόμενοι από μια χώρα που είδαμε ένα πραξικόπημα να ε, ε, δίνει ένα τέλος στην δικτατορία. Αυτό που έχει σημασία για την, για την παγκόσμια κοινή γνώμη είναι το μήνυμα το οποίο θα αποστείλει η, Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά σε, στους πολίτες, στην όλη η δημοκρατική διαδικασία, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει την εκλογική διαδικασία ε, στην Αίγυπτο μόνο εάν είναι γενική και συμπεριλαμβάνει του όλους. Και θα πρέπει και η κυβέρνηση να είναι οικουμενική αν θέλετε λίγο πολύ, όλοι να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και θα ήθελα να καταλάβει ο κύριος Λεόν ποιες είναι οι δυνάμεις ε, που παίζουν γιατί οι σαλαφίστες η Νούρα έπαιξε τον ρόλο, έπαιξαν τον ρόλο τους υποστηρίζοντας ε, την στρατιωτικό, το στρατιωτικό πραξικόπημα αλλά τώρα στην ε, θέσπιση των νόμων και τα λοιπά τι ρόλο θα παίξουν πρέπει να υποστηρίξουμε μια δημοκρατική διαδικασία οι γυναίκες γίνονται σεβαστές, δεν γίνονται τις ημέρες μας. Και θα πρέπει να έχουν πλήρη δικαιώματα και θα πρέπει να έχουν ελευθερία ε, έκφρασης της γνώμης τους. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Γκράνμπερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και ευχαριστώ που έχω, όλους τους προσκεκλημένους μας. Μπορούμε να συζητήσουμε τι συνέβη στο παρελθόν ε, τις τελευταίες μέρες επί μακρόν. Το σημαντικό όμως να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον για τη δημοκρατία, για τις εκλογές. Πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι δεν μιλάμε για λογοκρισία ή αυθαίρετες συλλήψεις που ισχύουν αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι αυτά είναι ε, απαράδεκτα από οποιονδήποτε κατάσταση κατα, ε, καταλάβει την, αρχή της, την εξουσία. Ε, στην τον Ιούλιο, στις 24 Ιουλίου ε, θα γίνει αυτή η πιστεύω ότι μέχρι τότε έχουμε αρκετό χρόνο για να του πούμε ότι ή θα ακολουθήσετε τη σωστή κατεύθυνση και θα συνεχίσουμε ή αλλιώς ε, αν ακολουθήσετε λάθος δρόμο θα ε, υπάρχουν οι συνέπειες. Ε, πιστεύω ότι όλες οι χώρες θα πρέπει να αντιδράσουν στις 27, 27 τελικά. Θα πρέπει να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα ότι θα πρέπει να υποφεληθούν από αυτές τις 15 μέρες για να λάβουν τις σωστές αποφάσεις. Τώρα για την κλιμάκωση προφανώς είναι πολύ πιο περιπλοκά τα πράγματα από μια θρησκευτική συμμετοχή πίστη αν θέλετε ή όχι. Δεν θα πρέπει να ζητάμε απλώς και μόνο όλοι να πάρουν μέρος. Πρέπει να δούμε πώς θα επιτρέψουμε σε όλους να πάρουν μέρος. Πώς θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση να ε, συγκαλέσει μια γενική συνδιάσκεψη, μια παγκόσμια συνδιάσκεψη που θα συμμετέχουν όλοι. Μπορούμε να το κάνουν. Μήπως ε, θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε και με άλλους Σαουδική Αραβία, Κατάρ για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Η κυρία Νέτσι είναι η επόμενη ομιλήτρια. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τη συμμετοχή τους σε αυτή τη συζήτηση. Θυμάμαι ότι παλαιότερα, συζητώντας για την Αίγυπτο, είχα προειδοποιήσει επανειλημμένος για αυτό που ονομάζω εγώ σενάριο αλγερινού τύπου, όπου η εκλογική διαδικασία διακόπτεται διότι το αποτέλεσμα των εκλογών δεν ευχαριστεί ιδιαίτερα τον πληθυσμό ή τη διεθνή κοινότητα. Φοβάμαι ότι εδώ είμαστε μάρτυρες μιας ε, παραλλαγής ενός τέτοιου σενάριου αλγερινού και είναι ιδιαίτερα ανησυχητική η κατάσταση διότι το πρώτο ερώτημα είναι τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε ε, την έκρηξη ενός εμφυλίου πολέμου. Εάν, ε, όταν τα κόμματα έρχονται σε ενοπλή αντιπαράθεση με το στρατό, αυτό είναι αιτία πολέμου. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη μας ανησυχία. Το κατά πόσο αυτό προτείνει η κυρία Μπράτνερ θα μπορούσε να παίξει κάποιο ρόλο. Δεν ξέρω. Οτιδήποτε μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο πρέπει να χρησιμοποιηθεί Πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα και ίσως και θα πρέπει να αναστείλουμε τη χρηματική ενίσχυση μέχρι να είμαστε βέβαιοι ότι η διαδικασία βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να επανέλθουμε σε αυτή τη συζήτηση και ειδικότερα στην έκθεση των ελεγκτών, η οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και που ναι μεν λέει ότι δεν είναι πολιτική, αλλά είναι πολιτική σε μεγάλο βαθμό και θα πρέπει να τη συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο επόμενο ομιλητή είναι ο κύριο Τάνοκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ μίλησα στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο επί του θέματος. Είμαι υπέρ τη στρατιωτική παρέμβαση στην Αίγυπτο ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω αιματοχυσία και χάος εμφύλιος πόλεμος. Και ως απάντηση στη δύναμη του λαού που απορρίπτει τη Μόρση και την κυβέρνησή του και τις προσπαθίες του να καταλάβει όλα τα επίπεδα εξουσίας και να επιβάλλει μια θεοκρατία στην Αίγυπτο με διακρίσεις και διώξεις κατά της ε, χριστιανικής μειονότητας των κοπτών. Εγώ λοιπόν εκ μέρους ομάδας μου είμαστε απολύτως υπέρ της νέας μεταβατικής κυβέρνησης η οποία βέβαια θα πρέπει να παραμείνει στην εξουσία το λιγότερο δυνατό μέχρι να μπορέσουν να λαβούν χώρα δημοκρατικές εκλογές για ένα νέο κοινοβούλιο και ένα νέο πρόεδρο. Έχουν γίνει πολλές συλλήψεις, Φρανσέσκα Μπαρατνέρ, και η ερώτησή μου είναι σε ποιο βαθμό αυτές αποσκοπούν σε νόμιμη ασφάλεια ή ανταποκρίνονται σε καθαρά εκδικητικές διαθέσεις της νέας κυβέρνησης. Πώς αξιοποιεί η Κομισιόν το γεγονό ότι η Αίγυπτο μπορεί να αποτελέσει φορά έδαφο τώρα για του τζιχαντιστέ από οπουδήποτε, από τη Συρία, τη Λιβύη, οπουδήποτε, σε μια προσπάθεια αποσταθεροποίηση αυτή τη χώρα με ένοπλη τρομοκρατική αντίσταση. Ευχαριστούμε κύριε Τάνοκ. Η κυρία Λέζινγκ, έχετε το λόγο. Σε ευχαριστώ πολύ. Συμμερίζω με τις απόψεις ότι δεν μπορούμε ισοπεδωτικά να κάνουμε λόγο για στρατιωτικό πραξικόπημα Παρ' όλα αυτά θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν προοδευτικές στάσεις ε, στο στρατιώ ε, ταυτόχρονα και ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις κατά το παρελθόν συνεργάστηκαν με τους μουσουλμάνους αδερφούς για να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο μέλλον λοιπόν με αυτούς. Ε, υπάρχουν και ξεχωριστές πολιτικές απαιτήσει για την εξουσία από πλευρά των στρατιωτικών. Αν την πολιτική αυτή εξέλιξη στην Αίγυπτο θέλουμε να την παρακολουθήσουμε και να την υποστηρίξουμε πολιτικά, πρέπει να μεριμνήσουμε οι απαιτήσει, τα αιτήματα του πληθυσμού, του λαού να ικανοποιηθούν. Υπάρχει ένα ευρύτατο κίνημα για περισσότερη και μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη, πολιτισμική ελευθερία, πολιτιστική ελευθερία και παρόμοια αιτήματα. Πρέπει να δούμε λοιπόν μήπως είχαν ε, αξιολογηθεί εντελώς ε, λάθος οι αδελφοί μουσουλμάνοι. Είχε ε, πάει και σε επίσκεψη στη Γερμανία, στη Μέρκελ ο, ο, κύριος Μόρση και σε σχέση με ε, με την ε, ε, σύλληψη και βασανιστήρια στην Αίγυπτο είχε πει πρέπει να υπάρξει μια νέα προσέγγιση. Ήταν τελείως λανθασμένη αυτή η προσέγγιση σε σχέση με την Αίγυπτο. Πρέπει να παρακολουθήσουμε τον πληθυσμό, το λαό και τα αιτήματά του και τις απαιτήσει του. Υπάρχουν εδώ και τοποθετήσεις όσον αφορά δεκάδες εκπροσώπους της πολιτισ... της... του κινήματος που είχαν συμμετάσχει σε αυτό το επαναστατικό κίνημα. Να λάβουμε σοβαρά υπόψη τα αιτήματά τους και τις απαιτήσει τους. Ευχαριστώ. Παντσέρι. Σας ευχαριστώ. Παντσέρι έχει τον λόγο τώρα. Ευχαριστώ. Πρέπει να σας πω με κάθε ειλικρίνη ότι θα μου άρεσε να ακούω από καιρό καιρό μια ανάλυση, μια ε, παρουσίαση λογική, ορθολογική ε, από κάποιον που ασχολείται ε, με αυτά τα οποία γίνονται στην Αίγυπτο, χωρίς να περνάμε από μία φάση σε μία άλλη, χωρίς να σκεφτόμαστε ε, κάναμε ό,τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας και τον ρόλο, τον αρκετά αρνητικό όπως θεωρώ εγώ ρόλο που έπαιξαν οι Αμερικανοί τον τελευταίο καιρό. Δεν θα πρέπει απλώς και μόνο να έχουμε μια γραφειοκρατική παρουσίαση των ε, ερευνών και των μελετών ε, και των εκθέσεων που έχουμε κάνει για την Αίγυπτο. Αυτή η ανάλυση θα πρέπει να γίνει, διότι αλλιώς δεν θα καταλάβουμε τι συμβαίνει και τι πρέπει να γίνει. Εγώ θεωρώ ε, ότι οι συνέπειες του πραξικοπήματος τώρα εμφανίζονται και θα εμφανιστούν ακόμα πιο έντονα στο μέλλον. Και σημειώνω ότι αυτός ο οποίος θα κερδίσει από όλη αυτή την ιστορία δεν θα είναι αναγκαστικά οι αδελφοί μουσουλμάνοι, αλλά οι σαλαφιστές, οι οποίοι έχουν μια πολύ ε, συγκεκριμένη διαχείριση, την πολιτική διαχείριση των συνεπειών του πραξικοπήματος. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, πιέσουμε έτσι ώστε είτε να γίνει μία διαβούλευση επιτόπου άμεσα με μαζική ε, συμμετοχή μας και παρουσία μας ε, διότι θα πρέπει να μιλήσουμε με όλους και έχουμε μιλήσει με όλους από όλες τις πλευρές και θα πρέπει επίσης να έχουμε και συγκεκριμένους πόρους που θα πρέπει να ε, προσφέρουμε, διότι αλλιώς η οικονομική κρίση θα αλλάξει και θα ε, ε, διαφθείρει αν θέλετε τις, τις εκλογές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε την μεγαλύτερη μουσουλμανική χώρα μπροστά μας, μπροστά στην πόρτα μας, που οδηγείται σε αναρχία και θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ε, προχωρήσουμε. Δεν ξέρω, ε, ακούγονται διάφορα, μιλάμε για διάφορα σενάρια από την Αλγερία, Αλγερίας, Πορτογαλίας, Τουρκίας κτλ. Ε, θα βρεθούμε μπροστά σε μια κατάσταση που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Ανακαλύπτουμε τώρα εκ των υστέρων ότι οι αδελφοί μουσουλμάνοι είχαν μια την οποία δεν γνωρίζαμε και ανακαλύπτουμε μετά για τον Μόρση ότι ο στρατός έμεινε ε, κυρίακος του παιχνιδιού. Είχαμε επαφές εμείς με τον στρατό για να ξέρουμε τι είχε στο μυαλό του και ανακαλύπτουμε ότι η Αίγυπτος δεν είναι η Σουηδία όσον αφορά την δημοκρατία. Ε, ναι και κάποιοι ε, ε, ζητούν να επανέλθει, η να επανέλθει η στη συνταγματική τάξη. Συνταγματική τάξη πια στην Αίγυπτο. δεν νομίζω ότι αυτά τα οποία λέμε λειτουργούν σε ένα περιβάλλον σαν και αυτό της Αιγύπτου. θεωρία εντάξει, φορμαλισμός όσον αφορά τους δημοκρατικούς ασμούς επίσης. Όμως δεν πρόκειται να μας βοηθήσουν όλα αυτά για να, λύσουμε την, να επιλύσουμε την κρίση. Και αυτό που μας είπε και το ελεκτικό συνέδριο είναι ακριβώς αυτό, ότι υπάρχει μια βοήθεια πολιτική και οικονομική, η οποία είναι πολύ φορμαλιστική και που συνδέεται με, τους, με, τα, με θεσμικά όργανα τα οποία είναι στην περιοχή και ε, βλέπουμε το αποτέλεσμα. Έχουμε απομακρυνθεί από την πραγματικότητα των Αιγυπτίων και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλήσει σε όλους. Έχουμε μιλήσει σε όλους, όχι βλέποντας πώς αντιδρούμε στις δυνάμεις ε, που εμφανίζονται τώρα ε, στην, ε, στην Αίγυπτο, οφείλω να ομολογήσω ότι συμμερίζομαι κάπως τον ρεαλισμό του συναδέλφου του κ. Τάνοκ και ίσως το πραξικόπημα να είναι πιο, να είναι καλύτερο, να είναι προτιμητέο από κάποια άλλη λύση. Έστω και αν ο στρατός δεν πρέπει να κρατήσει την εξουσία. Να σας υπενθυμίσω ότι η διερμηνία θα έχουμε μέχρι τις 12 και 40. Μετά θα χρειαστεί να συνεχίσουμε μιλώντας στα αγγλικά. κυρία Ρομέρο Λόπες. Σας ευχαριστώ. Πιστεύω ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την κατάσταση στην Αίγυπτο το πρώτο το οποίο θα πρέπει να πετύχουμε είναι η απόσυρση των στρατιωτικών από την εξουσία. Πραγματικά πώς θα μπορούσαμε να αποτρέψουμε αυτή η σύγκρουση να γίνει εμφύλιος πόλεμος. Δεν είναι το ίδιο μια σύγχυση, μια σύγκρουση με κάποια, κάποια θύματα, θύματα με μια σύγκρουση με εκατοντάδε θύματα. Πώ μπορούμε να αποτρέψουμε λοιπόν μια τέτοια εμφύλια σύραξη. Πρέπει αυτό να κάνουμε πρώτο, αν είμαστε ικανοί να το κάνουμε. Το δεύτερο, ω ικανότητα που θα έπρεπε να μπορέσουμε να αποδείξουμε, μακάρι να είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό, να είμαστε σε θέση να μπορέσουμε να ε, θέσουμε αυτού που βρίσκονται σε διαφωνία να συμφωνήσουν, να διαβουλευθούν. Μουσουλμάνοι Μουσουλμάνοι αδερφοί, σαλαφίστες, αντιπολίτευση να μπορέσουν συνεκτικά να δράσουν ώστε να υπάρξει μια μεταβατική κυβέρνηση, μια μεταβατική περίοδος. Πρέπει να γεμίσει, να πληρωθεί εντός εισαγωγικών με πολιτικό αντίκρισμα και όχι εν κενό σε σύγκρουση. Θα πρέπει έτσι να προαχθεί αυτή η προσπάθεια, να υπάρξει μια τέτοια ε, συμφιλίωση. Αυτή μπορεί να είναι η δική μας συνεισφορά. Πολιτική διαδικασία υπό τους όρους να προχωρήσει λοιπόν, να δώσουμε συνδρομή μας ώστε να υπάρξει αυτή η συνάφεια και συνεκτικότητα που σήμερα δεν υπάρχει. Διότι διαφορετικά θα έχει κάθε δικαιολογία το στράτευμα να παραμείνει στην εξουσία. Ευχαριστώ. Αρλάκη. Αρλάκη, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εκτίμησα ιδιαίτερα την επιφυλακτική θέση του Μπερναρντίνο Λεόν όσον αφορά τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κρίση. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Αραβική Άνοιξη μόλις ξεκίνησε. Θα είναι μια μακροχρόνια διαδικασία με πολλά σκαμπανεβάσματα και πολλά παράδοξα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι για αυτό το μακροχρόνιο χαρακτήρα της. Να μην πιστεύουμε ότι θα σταθεροποιηθούν τα πράγματα άμεσα. Και ποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι η δυναμική οι δυνάμεις ε, της Αιγύπτου, οι στρατιωτικές θα έρχονταν κατά ενός Ισλαμιστικού καθεστώτος. Ήταν λάθος να υποστηρίξουμε το όμως και το την μπορεί να σταθεροποιούσε την Αίγυπτο. Αυτό το λάθος που έκαναν ιδιαίτερα οι Αμερικάνοι δεν πρέπει να επαναληφθεί. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε μακροχρόνια οικοδόμηση θεσμών και οικονομική ανάκαμψη. Αυτή τη στιγμή θα ήταν εντελώ λάθος να μιλάμε για αναστολή της ενίσχυσης, της στήριξής μας προς την Αίγυπτο, διότι η όξυνση της οικονομικής κρίσης μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικά αποτελέσματα. Οι ΗΠΑ επίσης έκαναν το λάθος να μην μετατρέψουν τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια που δίνουν σε αρρωγή προς τους πολίτες. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια στρατηγική το να μην εμπλεκόμαστε υπερβολικά στις λεπτομέρειες της κρίσης, να διαβουλευόμαστε για την οικοδόμηση θεσμών. Ευχαριστώ. Thank you, Chairman. Επόμενη μιλήτρια, η κυρία Κρόμπεργκ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πολλά... Ένα ευρύτερο ερώτημα τίθεται στην Αίγυπτο αφορά την αξιοπιστία της δικής μας διαδικασίας υπεράσπισης της δημοκρατίας. Το ερώτημα είναι, μπορεί ποτέ να είναι ε, δημοκρατικό ένα πραξικόπημα. Μπορούμε να παραβλέψουμε τις ανησυχίες ε, αυτές του κατά πόσο οδηγείται προς δημοκρατία. Μπορούμε να παραβλέψουμε τις επιθυμίες των ανθρώπων που έχουν κατέβει στους δρόμους και κατά πόσο υποστηρίζουν αυτό το στρατό και κατά πόσο τον υποστηρίζουν οι ανθρωπιστικέ οργανώσει. Πιστεύω ότι υπάρχουν και κάποιε περιφερειακέ πτυχέ που θα πρέπει να σκεφτούμε. Πώ θα αντιληφθεί η Μέση Ανατολή τη δημοκρατία, αν αφορούσε το ζήτημα μόνο τη βία, το μέλλον, την οικονομία, τότε ο τρόπο που εμεί προσπαθούμε να υπερασπίσουμε τη δημοκρατία δεν θα φέρει αποτελέσματα. Πρέπει να είμαστε ε, αξιόπιστοι, να γίνουμε πιστικοί. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής, ο ε, κύριος Σόουετ. Παρακαλώ, ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αν θεωρήσουμε ότι η Αίγυπτος είναι ε, ένα πείραμα για τη δική μας εξωτερική πολιτική, ε, αυτή την ερώτηση πρέπει να κάνουμε στον κύριο Λεόν. Το είχαμε προβλέψει αυτό. Μιλούσαμε και πριν στους ανθρώπους, τους μιλάμε και τώρα. Πρέπει να δούμε τι ρόλο θα παίξουμε εμείς. Δεν έχουμε ευθύνη για το τι συμβαίνει αλλά πρέπει να καταλάβουμε κατά πόσο είχαμε αντιληφθεί τι γινόταν εκ των προτέρων και όταν λέτε να μην μας χρησιμοποιήσουν, ναι συμφωνώ, αλλά ποιος είναι ο ρόλος μας τώρα, εμείς απλά καθόμαστε και περιμένουμε. Θα ήθελα να ακούσω μια πιο θετική απάντηση εκ μέρους του κυρίου Λεόν για αυτό. Συμφωνώ με όλους όσους λένε ότι η κλιμάκωση είναι το πρώτο θέμα που μας ανησυχεί και στο οποίο πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα. Προς τους ομιλητές μας λοιπόν, αν αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε είναι ο εμφύλιος πόλεμος ε, όπου πολλοί θα χάσουν τη ζωή τους, τι κάνουμε γι' αυτό. Και τέλος, αν αιτιολογείται η στρατιωτική παρέμβαση και η άποψή μου είναι ίδια με τις συναδέλφους μου της κυρίας Γκόμες, η μόνη αιτιολόγηση θα μπορούσε να είναι το παρελθόν του καθεστώτος Μόρση που προωθούσε μια αντιδημοκρατική προσέγγιση. Συμφωνώ ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να κρίνει κατά πόσο ήταν σωστό ή λάθος το πραξικόπημα, αλλά πιστεύω ότι θα θέλαμε να ακούσουμε μια απάντηση από τους ομιλητές εδώ. Ευχαριστούμε. Αγαπητοί ομιλητές, έχετε 15 λεπτά για απαντήσεις. 5 λεπτά ο καθένας. Yes, Mr. Leon, you're the first. Well, thank you, thank you very much.